Good morning everybody. Καλή σας, α, καλή σας μέρα. Συζητήσαμε για το 2016. Μπάρμπαρα Ματέρα δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα που είναι η συγκήτριά μας ε, για την ε, έκθεση που πρέπει να συζητήσουμε τώρα που είναι ο προπολογισμός του 2016. Έχει αντικαταστάτη όμως. Η προθεσμία είναι 18 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Οπότε, η κυρία Σόντροβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η κυρία Ματέρα ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Εγώ ευχαρίστως να διαβάσω το σημείωμα που μου έδωσε. Η εμπειρία μας διδάσκει ότι όταν πρόκειται για τις γυναίκες στις διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού είναι πολύ δύσκολο να περάσουν στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Γι' αυτό λοιπόν στη γνωμοδότησή της η κυρία Ματέρα αναφέρει την άποψη ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάγκη ενσωμάτωση στοιχείων που έχουν να κάνουν με το φύλλο στις διάφορες διαδικασίες και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Βάσει της εμπειρίας που έχουμε μέχρι τώρα, η στρατηγική τι κάνει, συγκεντρώνει τα αιτήματα για τα πιο σημαντικά ζητήματα όπως είναι η βία, οι διαφορές στους μισθούς, οι πολιτικές για τις συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Αντί να ζητάμε υπερβολικά πολλά και να παίρνουμε τίποτα, να επικεντρωνόμαστε λοιπόν στα βασικά. Όπως ήδη ακούσαμε χτες κατά την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε για τον προπολογισμό 2016 με τον εισηγητή τον κύριο Φερνάντες, ε, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πέντε ζητήματα που ζητάμε από την Επιτροπή Προπολογισμών. Πρώτον, να διατηρηθεί το όνομα Δάφνη όσον αφορά τους συγκεκριμένους στόχους που έχουμε για να καταπολεμήσουμε την βία κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών. Δεύτερον, να χρησιμοποιούμε τη, τα κονδύλια του προπολογισμού ως αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόθεση της ισότητας των δύο φύλων. Τρίτον, να υπάρχει χρηματοδότηση στα προγράμματα τα οποία στηρίζουν και προωθούν την επιχειρηματικότητα των γυναικών, ιδιαίτερα στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρών και μεσαίων, στα επιχειρηματικά προγράμματα και στο κοινωνικό ευρωπαϊκό ταμείο. Τέταρτον, να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό κέντρο ελέγχου στα πλαίσια εκείνου που ήδη υπάρχει και να αυξηθεί το προσωπικό κατά μία μονάδα. Θεωρούμε ότι ο προπολογισμό του κέντρου αυτού πρέπει να παραμείνει. Πέμπτον, να υπογραμμίσουμε την αναγκαιότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα καταπολεμούν τα στερεότυπα που υπάρχουν σήμερα σε σχέση με τους άντρες και τις γυναίκες και θα προωθήσουν τις ίσες ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση και στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Sin. Αν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ να έρθετε σε επαφή με την κυρία Ματέρα και τη, τους συνεργάτες της, οι οποίοι θα σας απαντήσουν σε ό,τι απορίες ή σχόλια έχετε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σόντροβα. Τώρα, εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, οι σκιώδες εισηγητές, η κυρία Μπορσάν εκ μέρους των σοσιαλιστών έχει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία και όλους τους συναδέλφους για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία που προτάθηκε. Τα περισσότερα από τα προγράμματα που προτείνονται έχουν στόχους στη χειραφέτηση των, γυναικών, την οικονομική του ισότητα, την ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων, ώστε να μπορέσουν να εξισορροπήσουν τις ε, οικογενειακές, ιδιωτικές και επαγγελματικές τους ζωές. Ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο σήμερα, ειδικότερα σε χώρες που δεν ε, παρέχουν επαρκή υποστήριξη σε θέματα φροντίδας των παιδιών καθώς οι γυναίκες ε, πρέπει να φερώσουν χρόνο στη σταδιοδρομία τους. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η συστηματική ε, εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων και ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων ώστε να, οι γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα να είναι επιτυχείς επαγγελματίες και μητέρες. Είναι μακρύς ο δρόμος μπροστά μας, αλλά αν συνεργαστούμε μπορούμε να επιτύχουμε κάτι. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Βάινα, εκ μέρου των Πρασίνων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ επίσης και την εισηγήτρια για την υποβολή της γνωμοδοτήσεως που τη βρίσκω σωστή και η δική μου πολιτική ομάδα δηλαδή. Ένα από τα κεντρικά σημεία αναφέρεται και στην βία κατά των γυναικών. Το είπατε και εσείς προηγουμένως στη δήλωσή σας ε, είναι σημαντικό που το περιλαμβάνουμε στη γνωμοδότηση, συμφωνώ απόλυτα, αλλά θέλω να τονίσω ότι ο αγώνας κατά της βίας κατά γυναικών και παιδιών δεν μπορεί να θεωρηθεί μοναχά σαν αποστολή της ε, Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών. Είναι ένα καθήκον ολόκληρης της κοινωνίας. Βεβαίως είναι και σημαντικό και η ίδια η Επιτροπή Γυναικών να τοποθετηθεί. Έχουμε κάποιες ε, τροπολογίες βέβαια γιατί βρίσκουμε κάποιες ελλείψεις ή πάντως ορισμένα πράγματα πρέπει να ενισχυθούν. Το ένα είναι να τονιστεί η σημασία του κοινοτικού προϋπολογισμού για την ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής ε, θέσης των γυναικών. Μιλήσαμε χθε με τον κύριο Φερνάντες για τη Επιτροπή Προπολογισμών, δηλαδή που έχει υποβάλει σχετικέ κατευθυντήριε γραμμέ και όπου στοχεύει καθαρά στην χρήση και στη σημασία του κοινοτικού προϋπολογισμού για θέματα κοινωνικής συνοχής. Και από την Επιτροπή μας λοιπόν είναι σημαντικό να τονιστεί ξανά ο τομέας αυτός και ιδίως το ζήτημα του χάσματος των αμοιβών ε, μεταξύ των δύο φύλων. Gender Pay Gap που βέβαια τονίζεται ακόμα περισσότερο λόγω της κρίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί με προγράμματα και μέτρα. Το ίδιο για την δημιουργία απασχόλησης και μάλιστα πράσινων θέσεων απασχόληση. Και αυτό λοιπόν μπορεί να περιληφθεί εδώ. Επίσης το άρθρο 2 του, να, να εμφανίζεται το κοινωνικό ταμείο και η απασχόληση, μάλλον η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Αυτά πρέπει να επεκταθούν για να περάσουν σε όλα τα διαφθορτικά ταμεία, όλα τα διαφθορτικά προγράμματα και το Ταμείο της Αντιμετώπισης Παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή αυτό, αυτή η gender dimension, η πτυχή δηλαδή της ισότητας των φύλων πρέπει να περιληφθεί σε όλα αυτά. Για την πρόθεση των γυναικών στην επιχείρηση θέλουμε να αναφερθεί και η διευκόλυνση πρόσβασης σε μικροχρηματοδότηση, microfinancing δηλαδή. Ε, δηλαδή πρόσβαση σε πιστώσεις εν τέλει, θυμούμε ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα που είχε προωθήσει στη Γερμανία η Ευρωπαϊκή Ένωση προετών και που το έλεγαν τράπεζα γυναικών και που διευκόλυνε την πρόσβαση γυναικών σε πιστώσεις. Και αυτό νομίζω λοιπόν ότι θα είναι καλό να περιληφθεί ως πρωτοβουλία στη γνωμόδοτησή μας. Τέλος δε, όπως είπα και χθε στη συζήτηση με τον Φερνάντες, αυτό βέβαια συζητήθηκε ήδη δύο φορές, αλλά ως πυρήνας στην γνωμοδότησή μας να πει το gender budgeting, προτείνοντας και μεθόδους εφαρμογής του. Και όχι μόνο μια γενική μνήμα στην γνωμοδότηση, δηλαδή μια προτροπή να χρησιμοποιηθεί το gender budgeting όσο γίνεται περισσότερο. Ήδη πέρσι είχε εκδοθεί γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών με μια τροπολογία που πρότεινε μια μεθοδολογική προσέγγιση και θα έλεγα αυτήν την τροπολογία να την περιλάβουμε ξανά φέτο. Πάντω ευχαριστώ πολύ για την υποβολή τη νομοδοτήσεω, την οποία βρίσκουμε καταρχήν σωστή και χαίρομαι πολύ που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και άλλο για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βάνα. Άλλο κανεί. Εσεί κύριε Βιώ. Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Συμφωνώ με πολλά από όσα έχουν συμπεριληφθεί στη γνωμοδότηση το να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τη βία κατά των γυναικών να δούμε το EIGE και το, την ένταξη της διαστάσης του φίλου στον προεπολογισμό. που συζητήσαμε και χθε στην Επιτροπή Προεπολογισμών. Ε, είναι πολλά ήδη και πρέπει να ε, πιέσουμε για την ένταξη της διάθεσης του φίλου στον προπολογισμό. Τα χρήματα είναι ίσως ε, ένας από τους καλύτερους τρόπους ε, για να ενθαρρύνουμε δράση, οπότε δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά μετροπαθείς. Πρέπει να στοχεύσουμε ε, τις μικρές επιχειρήσεις και να δώσουμε στις γυναίκες την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας. Πρέπει λοιπόν να δοθούν ε, ευκαιρίες. Ε, δεν πρέπει να πούμε «Α σας παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και εντάξει και τη διάσταση του φίλου στον προπολογισμό». Όχι, πρέπει να υπάρχει ένα διευθυντικό ταμείο το οποίο θα διαθέσει πόρους ώστε να εξασφαλιστεί η ισότητα. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο για παράδειγμα μπορεί να επενδύσει για φροντίδα των παιδιών και για φροντίδα των ηλικιωμένων, και αυτό είναι ένα από τα σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να τονίσουμε από πλευρά μα. Όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών, εδώ ουσιαστικά αναφερόμαστε σε οικονομική εξάρτηση και χρειαζόμαστε ισχυρή, ισχυρό κράτος ε, ε, πρόνοιας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι, να μου διευκρινίσετε κάτι, γι' αυτό ζήτησα τον λόγο. Ε, αληθεύει και οι συνάδελφοι να το γνωρίζουν ότι από φέτο αλλάζει ο τρόπο που συζητάμε τον προπολογισμό. Εξ ολοκλήρω, ο κύριο Φερνάντε ε, μα ενημέρωσε σχετικά, όπω γνωρίζετε, ήδη. και ε, εγώ τώρα ως ε, μέλος της Συντακτικής Επιτροπής ε, για αυτή την έκθεση σε μια άλλη επιτροπή. Η έκθεση αυτή αποτελεί εντολή για τριμερή διάλογο, οπότε ο κύριος Φερνάντες θα μείνει πολύ ικανοποιημένος με αυτή την εντολή. Τρεις εκθέσεις προετοιμάζονται Ε, υπάρχουν τρία σημεία στα οποία εμεί ω Επιτροπή Γυναικών μπορούμε να έχουμε κάποια επιρροή, να πούμε πώ θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα και μετά να δούμε πώ θα ε, εφαρμοστούν ε, πρακτικά μετά. Έχουμε μια δεύτερη έκθεση όπου μιλάμε για κάποιε γραμμέ που θέλουμε να αλλάξουν. Τα πιλωτικά προγράμματα, για παράδειγμα. Τι ζητήματα εμεί θεωρούμε σημαντικά ω Επιτροπή Γυναικών. Δεν πρέπει να αναμειγνύουμε τα δύο διότι μιλάμε για συγκεκριμένα κονδύλια του προ... δεν μιλάμε ακόμα για συγκεκριμένα κονδύλια του προπολογισμού, μιλάμε για το ολοπλαίσιο, μιλάμε για την κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να κινηθεί. Με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε στην πρώτη έκθεση. Δεν είναι μεγάλη, είναι στοχευμένη και ασχολείται με θέματα που αφορούν την Επιτροπή μας και ε, αναφέρεται στην κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να κινηθούμε και ορίζει τις παραμέτρους. Ε, σε μεταγενέστερες εκθέσεις θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι θέλει να πάρει το λόγο, σωστά. Ναι, ευχαριστώ. Θέλω να πω κάτι τεχνικό βασικά για τη Δάφνη. Πρέπει να διευκρινίσουμε αυτό το σημείο. Η δημοσιονομική ονομασία έτσι όπως έχει σήμερα στον προϋπολογισμό βασίζεται στην νομική βάση του προγράμματος για την ισότητα και την ηθαγένεια. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις γραμμές στον προϋπολογισμό. Το θέμα που μας απασχολεί είναι το εξή. Έχουμε συγκεντρώσει τους εννέα ειδικούς στόχους του προγράμματος σε δύο διαφορετικές ομάδες. Και κάθε ομάδα αντιστοιχεί σε μία γραμμή του προπολογισμού. Αυτό εξηγεί την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Το πλεονέκτημα είναι η ευελιξία. Υπάρχει ευελιξία για τον κάθε ειδικό στόχο μέσα στην ίδια γραμμή του προπολογισμού. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στον ειδικό στόχο που αντιστοιχεί στη Δάφνη στο πρόγραμμα Statement. Έχετε το ποσό που και έχετε επίση και το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Εξάλλου, αν μέσω μιας τροπολογίας που προτείνει το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να προσθεθούν κονδύλια που αντιστοιχούν σε έναν ειδικό ιδιαίτερο στόχο, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φροντίσει για τα ποσά αυτά για το συγκεκριμένο ειδικό αυτό στόχο. Τέλος, όσον αφορά την προβολή, πρέπει να ξέρουμε ότι η ονομασία Δάφνη συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας. Είναι ενήμεροι οι διάφοροι παράγοντες και γνωρίζουν ότι προτείνουν προγράμματα για τη Δάφνη. Θέλω να πω κάτι και για το Ινστιτούτο για την Ισότητα μεταξύ των δύο Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τον εισηγητή για το ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τη βία σε σχέση με τα δύο φύλλα και ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών. Το Ινστιτούτο προετοιμάζει λοιπόν ένα στρατηγικό πλαίσιο για την βία κατά των γυναικών που θα καθορίζει προτερότητες και μεσοπρόθεσμους στόχους. Το τούτο λοιπόν μπορεί κάλλιστα να χρησιμεύσει ως κέντρο ελέγχου για την ε, βία ανάλογα με το φύλλο έτσι όπως προτείνει και η γνωμοδότησή σας. Η ενίσχυση τώρα μιας θέσης έτσι όπως το προτείνει η συγκήτρια σίγουρα θα οδηγήσει στον επιθυμητό στόχο, δηλαδή στη μείωση της βίας ε, σε βάρος των γυναικών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, τελείωσε η συζήτηση αυτή. Υπενθυμίζω την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, που είναι 8 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Περνάμε στην επόμενη συζήτηση, ενίσχυση της θέσης των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγήτρια είναι η κυρία Λιλιάν Ροντρίγε, η οποία θα μας παρουσιάσει την έκθεσή της και μετά θα συζητήσουμε. Παρακαλώ, η συγγήτρια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση για το θέμα αυτό. Συνέβαλαν σημαντικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως ε, τον κύριο Μαργάλ, τη Γραμματεία και ειδικότερα τον Μανουέλε και την Επιτροπή ΦΕΜ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον βρεθό μου που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συνταξία αυτού του εγγράφου. Πριν παρουσιάσω την έκθεση, ήθελα να μιλήσω για το κομμάτι που μιλάμε για τη χειραφέτηση των κοριτσιών μέσω της παιδείας. Εδώ πρέπει να κάνουμε τη διαφορά μεταξύ δύο διαφορετικών ενιών που ορίζουν, ε, κάνουν διακρίσεις και ε, συμπεριλαμβάνουν. Υπάρχουν δύο βασικοί στόχοι. Ο πρώτος είναι να διασφαλιστεί η χειραφέτηση των κοριτσιών μέσω της παιδείας και να είμαστε βέβαιοι ότι η σχετική συμφωνία υλοποιείται. Έχουμε διάφορου στόχου ε, να υπάρξει νοοτροπία σχολική για την ισότητα των φύλων. Δεύτερον, να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα σπουδών έχουν προσαρμοστεί ανάλογα. Τρίτος ε, συγκεκριμένος στόχος ε, να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων Στι ε, διαδικασίε λήψη αποφάσεων στον επαγγελματικό κόσμο, ειδικότερα όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση. Τέταρτος στόχος, αύξηση του ποσοστού συμμετοχή των γυναικών σε θέσει ευθύνη. Ε, πέμπτον, ε, διασφάλιση της οικονομική αυτονομία των κοριτσιών. Όσον αφορά τη μεθοδολογία μας, μελετήσαμε διάφορα ε, νομοθετήματα και χρησιμοποίησαμε δύο τεχνικές ε, αναλύοντας το περιεχόμενο. Καταλήξαμε σε έξι ευρείες κατηγορίες ε, ενημέρωση και προγράμματα σπουδών όχι μόνο στα σχολεία και στα σχέδια των σχολείων, στα προγραμματισμό των σχολείων, προγράμματα σπουδών γενικότερα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών συγκεκριμένα μέτρα. Μετά κοιτάξαμε την παρακολούθηση και την υλοποίηση προγραμμάτων και αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων. Επίσης ε, δημιουργήσαμε διάφορες υποκατηγορίες, σχολεία, θέσεις εργασία, μισθό. Δεν θα σας δώσω όλες τις πληροφορίες τώρα, ε, είμαι σίγουρο ε, ότι είστε όλοι εξοικειωμένοι. Αλλά θα ήθελα να περάσουμε στις συστάσεις γιατί επ' αυτών θα ψηφίσουμε ουσιαστικά, όχι επί των στοιχείων. Η έκθεση θεωρεί ότι η εκπαίδευση είναι στο μέσο που μπορεί να ενισχυθεί η θέση των κοριτσιών. Πρόκειται για κρατικού οργανισμού και έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν τι διακρίσει. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπω έχουν καταδείξει οι επιστημονικέ έρευνε, δεν παρέχουν απλά γνώσει. παρέχουν και κοινωνικές επεπιθήσεις και επεπιθήσεις περί φύλων. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία θα προωθούν την ισότητα σε όλα τα επίπεδα του σχολικού συστήματος, από το προνήπιο μέχρι το πανεπιστήμιο. Ε, η κατάρτιση του θέματος της ισότητας πρέπει, και για τους ε, διδάσκοντες ε, πρέπει να είναι συνεχής. Χρειάζεται να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων μεταξύ των ε, ε, διδασκόντων σε όλες τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης. Η ισότητα των φύλων πρέπει να αποτελεί κριτήριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών θα πρέπει να απαιτήσουμε την εισαγωγή του ίδιου προγράμματο σε σχολεία εθνικών μειονοτήτων και να παρέχεται ένα πρόγραμμα οικονομική αρρωγή ώστε να αποφεύγονται τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψη των σχολικών σπουδών που κυρίω αφορούν τα κορίτσια. Αυτά σύμφωνα με τι προτάσει του Συμβουλίου. Ένα άλλο βασικό κριτήριο, η κατάρτιση για τα προγράμματα σπουδών. Θεωρούμε ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στα προγράμματα σπουδών με επίσημο και ανεπίσημο τρόπο. Έχουμε τα επίσημα προγράμματα σπουδών και τα ανεπίσημα τα οποία συμπληρώνουν τα επίσημα. Και μετά υπάρχει κάτι για το οποίο μιλάμε ελάχιστα, τα κρυφά προγράμματα σπουδών, τα οποία ε, χρειάζονται περαιτέρω ε, παρέμβαση στην Ευρώπη. Πρόκειται για κοινωνικά ζητήματα, κοινωνικέ αξίες ε, που μεταβάζουμε στα παιδιά. Έχουμε λοιπόν το περιεχόμενο των προγραμμάτων, ε, τα σχολικά προγράμματα, ε, οι δραστηριότητες πέραν της παιδεία και οι αθλητικές δραστηριότητε είναι σημαντικές εδώ. Πρέπει να παρέχουμε πληροφορίες και να διασφαλίζουμε ίση πρόσβαση στις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής για αγόρια και κορίτσια από το προνήπιο. Μιλάμε εδώ για ε, γνώσεις ε, της ψηφιακής τεχνολογίας ώστε να αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις για τις επιστήμες, τη τεχνολογία και τις τεχνολογίες προφοριών και επικοινωνιών ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα δοθούν οι δυνατότητε σε κορυφαία να επιχειρηματίε. Σε συνεργασία λοιπόν με τι τοπικέ αρχέ πρέπει να διασφαλιστούν ε, τέτοιες, ε, ε υπαρχή τέτοιων γνώσεων μαζί με τι τοπικέ κοινότητε ε, και που φυσικά να περιλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου. Αυτό πρέπει, μπορεί να γίνει και με online μαθήματα. Οι εκδότες ε, σχολικού υλικού θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των κοριτσιών θα αποτελεί επίση κεντρικό ζήτημα κεντρικό θέμα. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι πληροφορίες περισσότερες των φίλων να αποστέλλονται και σε γονείς. ώστε να ε, άρουμε στερεότυπα τα οποία υπάρχουν ήδη. Εδώ μπορούμε να πιστεύουμε, ε, καθώς πιστεύουμε ότι ένας ε, δάσκαλος μπορεί να φέρει κοινωνική αλλαγή μπορεί να φέρει και την ενίσχυση της θέσης των κοριτσιών. Τώρα όσον αφορά τους εργοδότες, η ισότητα των φύλων στην παιδεία είναι σημαντική, αλλά όσοι εργάζονται με μικρά παιδιά και όσοι φροντίζουν παιδιά πρέπει να θεωρούν ε, ότι οι δουλειές τους είναι το ίδιο άξιος όσο οι κλασικές δουλειές ε, της αγοράς εργασίας. Όσον αφορά τις επενδύσεις, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των διαφορών πολιτικών ε, χρειαζόμαστε τις απαραίτητες αρχές όπως το Υπουργείο για παράδειγμα παιδείας με κάποιον ειδικό φορέα που να ασχολείται με την ισότητα των φύλων Πρέπει η ισότητα των φύλων να αποτελεί ε, βασικό κριτήριο αξιολόγηση ε, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και θα πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα αξιολόγηση μελλοντική νομοθεσία για τέτοια θέματα επίση. Και θα μπορούσε να υπάρχει ένα ετήσιο βραβείο ισότητα των φύλων ε, και να ρίχνουμε τα κράτη-μέλη για κάτι τέτοιο. Το τελευταίο που έχω να πω. Όλα αυτά θα κοστίσουν, αλλά μέσω του οριζόντα 2020 και ε, χάρη στην Ευρωπαϊκά Ταμεία λογικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ποιο θέλει το λόγο. Με κυρία Βέρδερ. Ευχαριστώ, καθώς επίσης ευχαριστώ και την κυρία Ροντρίγκες Φαίνεται σύντομη η έκθεση, αλλά έχει, είναι πλούσια σε περιεχόμενο. Και βεβαίω είναι περιεκτική. Περιλαμβάνει πολλά θέματα παιδεία και του ρόλου που μπορούμε να παίξουμε εμεί για να ενδυναμώσουμε, empower δηλαδή, τα κορίτσια και τι νέε γυναίκε. Και για εμά, ω Ευρωβουλή είναι μια ευκαιρία να τοποθετηθούμε σχετικά με τις προτεραιότητες παρόλο που βέβαια όπως και στην υγεία ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός και στην παιδεία. Τώρα αυτή η ενδυνάμωση μέσω της παιδείας έχει δύο σχέδια. Αφενός η ενδυνάμωση, η παιδεία μάλλον, ε, βοηθάει μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό τη συνοδεύει σε όλη τη ζωή τους. Και αν αρχίσει από νωρί, υπάρχει και η δυνατότητα να φτιάξουμε και μια πιο ίση κοινωνία. Δεύτερο και μεταξύ άλλων, η παιδεία επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να αυξήσει τις δυνατότητες απασχολησιμότητάς του. Και αφήσει αυτό είναι μακροπρόθεσμο. Και επομένως και εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα και ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όσον αφορά την εκπαίδευση, οι δάσκαλοι, το λέει και η έκθεση, έχουν μεγάλο, μεγάλη δυνατότητα να παρέμβουν. Και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντική και σωστά τα λέει η έκθεση και για την αρχική και για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και πολύ καλά κάνει η έκθεση και λέει ότι και μιλεί για αγόρια και κορίτσια κορίτσια και αγόρια γιατί συχνά οι δάσκαλοι λένε αγόρια και κορίτσια και αυτό βέβαια έμεσα υπόγεια μεταδίδει ένα μήνυμα Νομίζω επίσης ότι χρειαζόμαστε, χρειάζεται να ενισχύσουμε την ε, πρώιμη εκπαίδευση. Μια, οι χώρες μέλη πρέπει να κάνουν και περισσότερο έτσι ώστε να προσαρμόσουν και τη φρασιολογία τους εκπαιδευτική και να ενθαρρύνουν και κορίτσια και αγόρια να προχωρήσουν, να μορφωθούν και σε μη παραδοσιακούς τομείς των ε, σχολικών προγραμμάτων. Τα λέει καλά. Λοιπόν, η έκθεση και για την κατεύθυνση που λαμβάνουν τα κορίτσια στις, ε, στην εκπαίδευσή τους. Χρειάζεται λοιπόν εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, χρειάζεται πρότυπα ρόλων γυναικών, δηλαδή και επιστημόνισες να πάνε στα σχολεία και να ενθαρρύνουν και τα σχολεία να πάνε να επισκεφθούν τα επιστημονικά ιδρύματα και να βελτιωθεί και ο επαγγελματικό προσανατολισμός που συχνά είναι πολύ αδύναμος Επίσης πρέπει να κάνουμε πιο ανθρώπινη την επιστήμη. Συχνά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εμφανίζουν σε επιστήμονες σαν κάποιους ημίθεους που φοράνε λευκές ε, ποδιές και είναι πολύ απομακρυσμένοι από την κοινωνία. Υπάρχουν όμως τομείς όπου βέβαια τα κορίτσια εκπροσωπούνται περισσότερα και αυτό που γνωρίζω εγώ καλά το τομέα είναι primatology, δηλαδή είναι η επιστήμη που ασχολείται με τους ε, εφιέστερους των πυθίκων, δηλαδή ε, τους, ε, μοιάζουν περισσότερο με ανθρώπους. Και εκεί παίζουν πολύ έντονο, ε, πολύ σημαντικό ρόλο οι γυναίκες. Επίσης σημαντική είναι και η δραστηριότητα εκτός σχολείων. Είναι σημαντικό να περιληφθεί λοιπόν και αυτή η εξωσχολική δραστηριότητα στην έκθεση γιατί επιτρέπει και στα κορίτσια και στα αγόρια να ε, διαρευνούν νέους ρόλους. Υπάρχει βέβαια και ένα θέμα πόρων πάντοτε και αυτό σε όλη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να τονίσουμε και την ανάγκη να προστατευτούν οι πόροι αυτοί, καθώς επίσης και να βελτιωθεί η χρηματοδότηση. Και νομίζω ότι υπάρχει μάλιστα και μια κίνηση προς την κατεύθυνση της ε, παρουσίασης περισσότερο των γυναικών που συμμετέχουν σε αθλήματα και γυναικείων πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Θα πρέπει όμως να τονωθεί κάπως η παρουσίαση αυτών των ε, γυναικείων συμμετοχών στα αθλήματα. Τώρα το επιχειρήν, εκπαίδευση για το επιχειρήν. Αυτό ακροθυγώς μόνο αναφέρεται στην εκθεσή και πρέπει να τονωθεί, να τονιστεί. Γιατί οι επιχειρηματίες είναι αυτοί που δημιουργούν την απασχόληση της αύριο. Να ενθαρρυνθούν λοιπόν κορίτσια και αγόρια να προχωρήσουν και σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα με το επιχειρήν που συχνά συνδέεται με την ανάληψη κινδύνων. Ήδη το επιχειρήν αυτό σημαίνει. Οι γυναίκες και κορίτσια γενικά δεν χαίρονται τόσο να αναλαμβάνουν κινδύνους όπως οι άνδρες. Όταν μιλούμε για επιχειρήσεις που αρχίζουν τη δουλειά τους, startup, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Ίσως έτσι είναι καλύτερα να το πούμε γιατί τότε αισθάνονται οι γυναίκες πιο άνετα. Ας εξετάσουμε λοιπόν τη φρασιολογία που χρησιμοποιούμε και εκεί. Και τέλος ε, η εκπαίδευση για τις γενετήσιες σχέσεις και τα λοιπά. Σεξ και σχέσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιώδες για να αντιμετωπιστούν ευρύτατες ανισότητες βασισμένες στο φύλλο μεταξύ γυναικών και ανδρών. Να μάθουμε στα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν τα προφυλακτικά. Χρειάζεται αυτή η εκπαίδευση γιατί αυτό ενισχύει τα κορίτσια και τις κοπέλες να δουν το σώμα τους πιο σωστά. Ότι δεν είναι δηλαδή παθητική συμμέτοχη σε μια σχέση, αλλά ότι έχουν τη δυνατότητα, έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις που του απασχολεί. Και ε, θα πρέπει να γίνει και υποχρεωτική μάλιστα εκπαίδευση αυτή. Γυναίκες ή κορίτσια τα οποία έχουν αυτό το empowerment μπορούν ε, να πάρουν καλύτερες αποφάσεις στα ε, θέματα που τις αφορούν. Και τα βλέπουμε αυτά και καθημερινά και στα media και θα πρέπει να ενισχύσουμε τα κορίτσια και αυτός είναι ο παιδευτικό ρόλο που πρέπει να παίξουμε. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για το σχέδιο χθε και με υπομονησία μένω και τι άλλε τροπολογίε. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Πετήρη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό η σημασία της εκπαίδευσης και της εργασίας για τις γυναίκες να υπογραμμιστεί στην έκθεση αυτή. Είναι σημαντικό επίσης να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στις απασχολήσεις αυτές σε ηγετικές θέσεις και είναι σημαντικό να φεύγουν λιγότερες γυναίκες από το σχολείο, να υπάρχει επίσης η ψηφιακή τεχνολογία και στην Ήπεθρο και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις φιλετικές διακρίσεις, το σεξισμό. Η εκπαίδευση είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτή και οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να μπορούν να καταπολεμήσουν τα στερεότυπα όταν πρόκειται για τη δουλειά που θα διαλέξουν. Στην έκθεση αυτή βλέπω και κάποια προβληματικά σημεία. Είναι τα σημεία 11 και 12 τα οποία απευθεία ζητούν από τις γυναίκες και τα κορίτσια να δοκιμάσουν νέους ρόλους και να αλλάξουν μεταξύ τους ρόλους. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους ανθρώπους να διαλέξουν μια διαφορετική ταυτότητα, να αλλάξουν ρόλο και ταυτότητα σε σχέση με αυτή τη ταυτότητα με την οποία έχουν γεννηθεί. Οι διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών πρέπει να γίνονται σεβαστές. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, ότι έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις από τις οποίες ξεκινούν και ότι τα παιδιά ανεξαρτήτως φύλου πρέπει να έχουν εξίσου πρόσβαση στην εκπαίδευση και πρέπει να μπορούν να αναπτύξουν την ταυτότητά τους συμπληρωματικά με την ε, ταυτότητά τους ως άτομα διαφορετικού φύλου. Τα κορίτσια πρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες και δεν πρέπει να τους ζητάμε να διαγράψουν τις, διαγρα... διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο φύλων. Θα ήθελα να τα σκεφτούμε αυτά, κυρίως τα σημεία 10 και 11, διότι δεν πιστεύω ότι συνεισφέρουν στην παρετέρω ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι διαγράφουν αυτό το οποίο μας δίνει την ταυτότητά μας, μα λέει το ποιοι είμαστε. Ευχαριστούμε. Κυρία Πίρκ. Θα ήθελα. Ε, να μιλήσω ειδικά, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί η έκθεση αυτή είναι εξαίρετη. Ήδη από την αρχή η έκθεση αυτή επιμένει στη σημασία που έχει η εκπαίδευση αν θέλουμε πραγματικά να πάψει να υπάρχει αδικία. Στα σουηδικά δύσκολα μπορούμε να μεταφράσουμε τον αγγλικό όρο empowerment. Παρόλα αυτά είναι κάποιο είδου απελευθέρωση και αυτήν μπορεί να τη δώσει η εκπαίδευση. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό το κάθε παιδί να έχει 100 δυνατότητες και όχι μόνο μία και δύο. Δεν υπάρχουν μόνο δύο μοντέλα. Υπάρχουν τουλάχιστον 100 μοντέλα για το μέλλον του κάθε παιδιού. Το κάθε παιδί θα πρέπει να μπορεί να ονειρεύεται βάσει αυτών των 100 μοντέλων και να διαλέξει. Δεν μπορούμε να του ζητάμε να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο μοντέλα και τίποτα άλλο. Πιστεύω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή πολύ σωστά επιμένει και λέει ότι πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα όποια και αν είναι αυτά. Πολλά από αυτά που ήθελα να πω τα είπαν άλλοι. Όμως θέλω να υπογραμμίσω ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις μας είναι κάτι πολύ σημαντικό και επιτρέπει στα κορίτσια να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν τι θα κάνουν με το δικό τους το κορμί. Έχουν έτσι τη δυνατότητα να αντισταθούν στη βία. Στη Σουηδία έχουμε μαθήματα αυτοάμυνας για τα κορίτσια με μεγάλη επιτυχία. Έτσι μπορούν τα κορίτσια και οι γυναίκες να μάθουν καλύτερα να προστατεύονται, να μείνονται. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος των σχολείων. Είναι αλήθεια ότι έχουμε βάλει πολλές ελπίδες στα σχολεία, στους διδάσκοντες, είναι όμως σημαντικό γιατί χάρη στο σχολείο μπορεί να ενισχυθεί ο ισότιμος ρόλος ανδρών και γυναικών, κοριτσιών και αγοριών καταρχήν. Έπειτα, πέρα από τα όσα λέει η έκθεση αυτή, θα μπορούσαμε ίσως να επιμείνουμε περισσότερο και σε αυτό που είναι η απελευθέρωση, τι σημαίνει και έτσι φτάνουμε και στις θέσεις εξουσίας, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για τον επιστημονικό τομέα. Πρέπει να έχουμε περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις και στον επιστημονικό κόσμο. Αυτό ίσως θα μπορούσαμε να το υπογραμμίσουμε περισσότερο στην έκθεση. Θέλω να προσθέσω ακόμα ότι στην δουλειά μας, στη διεθνή σκηνή, απέναντι δηλαδή σε τρίτες χώρες, είναι σημαντικό να υπογραμμίζουμε τη σημασία που έχει η εκπαίδευση των γυναικών. Είναι σημαντικό για να αποφύγουμε έτσι τη σεξουαλική εκμετάλλευση, να αποφύγουμε την θνησιμότητα των ε, γυναικών που σε διάφορα μέρη του κόσμου πεθαίνουν κατά τη γένα. Όλα αυτά είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με την δικιά μας αναπτυξιακή πολιτική. Το θέμα του φίλου είναι κάτι που πρέπει να εισαγάγεται τα σχολικά προγράμματα. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Καλπέτη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πριν πω την άποψή μου ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Θα ήθελα να μάθω κατά πόσο σύμφωνα με τον κανονισμό πότε μπορούν οι σκιώδεις εισηγητές να πούν τις απόψεις τους γιατί είμαι νέο μέλος στην ΕΚΟΝ και στην ΕΜΚΟ είμαι νέο μέλος εδώ και στην ΕΚΟΝ και στην ΕΜΚΟ έχουμε πολύ σαφείς κανόνες πρώτα απ' όλα εκφράζουν τις απόψεις τους οι σκιώδεις εισηγητές και δεν χρειάζεται να πούν ότι θέλουν τον λόγο, παίρνουν τον λόγο αυτόματα. Οπότε ήθελα να ρωτήσω σύμφωνα με τον κανονισμό πώ λειτουργούν τα πράγματα σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Pues miren, Κοιτάξτε. Είπαμε οι σκιώδεις καταρχήν, αλλά έχω εδώ διάφορα ονόματα και έτσι καλλιώς τέσσερις είμαστε εδώ, πέντε θέλουν όλοι να πάρουν το λόγο, θα πάρουν όλοι το λόγο. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ σημασία πόσο. Εδώ έχουμε γράψει τα ονόματα έτσι όπως με τη σειρά με την οποία εκδηλώσατε ενδιαφέρον. Απλά ρωτούσα για τους κανόνες. Μπορείτε να απαντήσετε αυτό που ρώτησα. Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες στην Επιτροπή μας για τη σειρά με την οποία παίρνουν το λόγο οι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πολύ. τότε θα δηλώνω ότι θέλω να μιλήσω στο μέλλον. Λοιπόν, ήθελα να πω την απόψη μου για ένα πολύ σημαντικό θέμα Είμαι πεπισμένη ότι θα αποτελούσε, έχουμε ένα εξαιρετικό τίτλο στην έκθεση αυτή, οπότε θα ήθελα να είναι εξαιρετική και η έκθεση. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Ε, είναι καταρτισμένη στο θέμα αυτό και αναφέρεται σε πολύ σημαντικά θέματα. Μιλάμε για το ρόλο που παίζουν οι γυναίκες και προσπαθούμε να πάμε πέρα από το απλά να αναφέρουμε το θέμα αυτό στην ημέρα των γυναικών. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι έχουμε ένα κοινό στόχο. Πρέπει να διασφαλίσουμε παιδεία υψηλού επίπεδου σε όλα τα δυνατά επίπεδα και πρέπει να διασφαλίζουμε πρόσβαση σε τέτοια παιδεία υψηλού επίπεδου για τα κορίτσια και για τις γυναίκες. Αναφερόμαστε στη σπουδαιότητα της παιδείας και της εκπαίδευσης ε, έκτακτα περιστατικά επίσης, σε, σε δύσκολες ε, ε, καταστάσεις. Μια σωστή κοινωνία θα οικοδομηθεί μόνο εφόσον να ενσωματώσουμε το κατάλληλο περιεχόμενο στα εκπαιδευτικά συστήματα. Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όχι μόνο διότι βοηθά τους ανθρώπους να επιτυγχάνουν και να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητές τους, επιτρέποντας τους να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, αλλά επίσης επειδή μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας. Όταν κάποιος μορφωθεί, μπορεί να ξεφύγει πιο εύκολα από τη φτώχεια. Αυτό χρησιμεύει επίσης και για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας. Ε, κάτι που θα επιτρέψει στα κορίτσια και στις γυναίκες να διαδραματίσουν ε, ε, πιο κέριο ρόλο. Είμαι επίση πεπισμένη ότι όταν μιλάμε για την εκπαίδευση των κοριτσιών, ένας από του καλύτερου τρόπου να ε, επιτευχθεί κέρδος από επένδυση είναι το να επενδύσει κανείς τα κορίτσια, διότι είναι μια αναξιοποίητη πηγή δυνατοτήτων. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους που πρέπει να συμπεριλάβουμε στην έκθεση είναι για παράδειγμα η εκπαίδευση ε, διδασκόντων ε, ανώτατης εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμού ώστε τα κορίτσια να μπορούν να αποκτούν τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες. Επίσης δίνει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην καταπολέμηση των στερεότυπων. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Διότι ξέρετε εμένα το πρώτο μου πτυχίο αφορά, είναι σε τεχνικό τομέα πληροφορική και έχω και διδακτορικό σε ένα παρόμοιο θέμα. Οπότε είμαι πεπισμένη ότι όσοι θεωρούν ότι πρέπει να ε, βοηθήσουμε τα κορίτσια για να αποκτήσουν περισσότερο θάρρος έχουν δίκιο. Μόνο εμείς μπορούμε να φροντίσουμε να υπάρχει το απαραίτητο πλαίσιο για να το βοηθήσουμε και η ψηφιακή διάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όταν μιλάμε για τον τομέα της πληροφορικής και ε, της επικοινωνίας, ε, τον ICT, πρέπει να βελτιώσουμε τα όσα προσφέρουμε εκεί. Άκουσα και σε προηγούμενους ομιλητές και συμφωνώ. Στην... Πρέπει να ε, περιοριστούμε στο θέμα της έκθεσης και να μην ε, ξεπεράσουμε τα ωραία του. Διαβάζοντας τις διάφορες παραγράφους που δεν είναι απόλυτα σαφείς, Θα μπορούσαμε σε περιπτώσει που δεν υπάρχουν σαφείς ορισμοί να κάνουμε παραπομπή σε σαφείς ορισμού. και κάποια θέματα έχουν αναμειχθεί εδώ πέρα, υπάρχει κάποια σύγχυση, οπότε θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε λίγο. Ίσως μπορούσα, θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε ορισμένα κομμάτια. Συμφωνώ ότι η παιδεία και τα σχολικά προγράμματα είναι πολύ σημαντικά. Εγώ είμαι μητέρα τριών, έχω δύο κορίτσια. Οπότε θεωρώ ότι αυτά που βλέπω εδώ στην έκθεση δεν είναι αρκετά. Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα διότι η αγορά δεν μπορεί να αξιολογεί τα κορίτσια βάσει αυτών. Είναι πολύ σημαντικό να τους προσφέρουμε ε, επαρκείς γνώση ώστε οι ικανότητες τους, τους οι δεξιότητές τους να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην εργασία τους. Μου είχαν πει εμένα τότε ότι δεν μπορούσα να γίνω μηχανικός και εγώ μου πεπισμένο ότι μπορούσα να γίνω μηχανικός. Οπότε θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια. Είναι καθήκον μας αυτό σε αυτόν τον τομέα. Είμαι βέβαιο ότι θα έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία. Όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα από το πλαίσιο της Διεθνούς Υμέρας για τις Γυναίκες. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η κυρία Σόιντεροβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτό το θέμα για την ενίσχυση θέση των κοριτσιών και την εκπαίδευσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό. Με την εκπαίδευση μπορούμε να επηρεάσουμε, μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Τα είπαμε, τα είπαν και οι συνάδελφοι πριν από μένα. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ένδια, για παράδειγμα, όπως είπε και η συνάδελφος. Όπως και εσείς, θέλω κι εγώ να ενθαρρύνω, να υποστηρίξω τα κορίτσια Θέλω όμως να παραμείνουν κορίτσια. Θέλω δηλαδή να διατηρήσουν την ταυτότητά τους ως κορίτσια. Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να παραμείνουν γυναίκες, ακόμα και αν υπάρχει ισότητα. Θέλουμε να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες τα κορίτσια όπως έχουν τα αγόρια, αυτό ναι. Θέλουμε να μπορούν και να συμμετέχουν και σε τομείς που θεωρούνται σήμερα περισσότερο αντρικοί στις επιστήμες, στο τεχνικό τομέα. Αλλά επαναλαμβάνω, στις, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στα πανεπιστήμια, είναι κυρίως κορίτσια που συμμετέχουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα, στα μάστερς είναι 50-60% γυναίκες που συμμετέχουν στα μάστερς. Η εκπαιδευτική πολιτική λοιπόν είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Είναι πολύ δύσκολο να επηρεάσουμε, να διακανονίσουμε εμείς τα προγράμματα τα εκπαιδευτικά των χωρών μελών. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε, να δώσουμε κίνητρα με οικονομικά προγράμματα κυρίως πιστεύω για να αλλάξουν κάπως τα προγράμματα και πώς να σας το πω αυτό ώστε να συμμετέχουν περισσότερο οι γυναίκες στους κλάδους που θεωρούνται περισσότερο για τα γόρια, τους τεχνικούς κλάδους για παράδειγμα. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που την αναφέραμε αρκετές φορές εδώ, όντως είναι μια ευκαιρία, αλλά είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτό το πιο σημαντικό στο θέμα που εξετάζουμε. Empowering ε, Girls, ενίσχυση της θέσης των κοριτσιών είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ είναι άλλα πράγματα που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Αυτά που είπαμε αλλά όχι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό το θέμα είναι πολύ ειδικό. Ε, μάλλον δεν είναι ότι φοβάμαι ότι είναι έτσι, είμαι σίγουρη ότι είναι έτσι και ότι είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Δεν θα ήθελα να συμπεριληφθεί στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος ευρωβουλευτής τον λόγο, εκτός αν ξεχνάω κάποιον. Τότε θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά η συγκήτρια πάλι. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά και καλωσορίζει την έκθεση αυτή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή αυτή για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Ε, εγώ αντικοστώ τον κύριο Αγκαλιανό, αλλά συνεργαστήκαμε τον κύριο Καλιάνο και έχουμε συνεργαστεί για πολύ καιρό μαζί επειδή πολλές φορές συμμετείχαμε ε, στη δουλειά αυτή και εκτιμάμε τη συνεργασία έχει συνοχή με τον τρίτο στόχο της, του πλαισίου ε, παιδείας και επαγγελματική κατάρτισης 2020 που ελαμβάνει την κοινωνική ένταξη, τις ευκαιρίες και την ηθαγένεια. Οπότε συνάδει όλο αυτό και συμφωνούμε και εμεί μετά όσα υπόθηκαν. Στο πλαίσιο αυτή τη δραστηριότητα, σημαντικό θα ήταν να υποθυμίσουμε στα κράτη-μέλη ότι μπορούν να κινητοποιήσουν σημαντικού πόρου από το ESIF για να βελτιώσουν την ισότητα των φύλων στον τομέα τη παιδεία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο ξανά στην εισηγήτρια για κάποια τελευταία λόγια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για όλα σας τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Ίσως κάποιοι τομείς που αγγίξαμε στην έκθεση δεν είναι σαφείς στα σημεία 11 και 12 που μιλάμε για τους κοινωνικούς ρόλους. Δεν αναφέρομαι εδώ στις παραδοσιακούς ε, ρόλους, ε, αναφέρομαι σε ρόλους ας πούμε ηγεσίας, ε, για να ενθαρρύνουμε την αίσθηση ηγεσία. Σε αυτή την έκθεση προσπαθούσαν να πω τα πράγματα λίγο στα γρήγορα, επειδή είναι μικρή έκθεση. Οπότε ίσω να μην ήμουν απόλυτα σαφή όταν αναφέρομαι σε νέου ρόλου στο σημείο 11. Μιλήσαμε, μιλάμε για την εκπαιδεία, ε, για τα σχολικά μαθήματα. Δεν μιλάω για γυναίκες ε, απαραίτητα που αναλαμβάνουν το ρόλο τους ως γυναίκες. Ε, μιλώ για ρόλους ηγεσία που είναι σημαντικοί στο πλαίσιο, σε ένα σχολικό πλαίσιο. Τώρα, για το ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης δεν παίζεται πιο σημαντικό ρόλο σε αυτή την έκθεση διότι ουσιαστικά εδώ κυρίως αναφερόμαστε την ε, σπουδαιότητα της ε, ενδυνάμωσης ε, των κοριτσιών στην παιδεία. Ξέρουμε διάφορα προγράμματα σπουδών μπορούν να θεωρηθούν ως κίνητρο για την ισότητα των φίλων. Δεν κατάλαβα την επίκριση που αφορούσε την εκπαίδευση ανθρώπων την εκπαίδευση ανθρώπων και κατά πόσο ε, ε, ε, επαρκώ αυτή την έκθεση. Δεν είμαι βέβαια αν κατάλαβα καλά. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Είπατε ότι δεν αναφέρομαι στην εκπαίδευση των διδασκόντων, αλλά την αναφέρω σε διάφορα σημεία τη έκθεση. Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για περισσότερες ε, συστάσεις. Θα προσπαθήσω να πλουστεύσω τη γλώσσα αλλά απέφυγα την επιστημονική γλώσσα όποτε μπορούσα. Αλλά όταν μιλάμε για την εκπαίδευση ως τρόπο ε, καταπολέμησης της φτώχειας, κάτι τέτοιο είναι σημαντικό. Λέμε ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε την ισότητα των φύλων και την ίση πρόσβαση Αναφέρθηκα στις κατηγορίες ε, που στην κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται στο παρελθόν. Είναι σημαντικό όταν μιλάμε για την πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών, την ίση πρόσβαση στην ε, παιδεία. Χρησιμοποίησα την ορολογία που χρησιμοποιούσαμε και στο παρελθόν. Δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι η παιδεία ως εργαλείο ε, καταπολέμησης των ανισοτήτων αναφέρεται μόνο στην επίσημη παιδεία. Εγώ μιλάω όμως και για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Στο σημείο 17 ε, πιστεύω ότι γίνεται πολύ ε, σαφές. Θα μπορούσαμε ίσως να, δώσουμε, να επισημάνουμε περισσότερο το ζήτημα της επιχειρηματικότητας. Χρήσιμο θα ήταν κάτι άλλο χρήσιμο που αναφέρεται επίσης στην έκθεση. Ενδεχομένως η σχέση με τα πρότυπα τα πρότυπα ανθρώπων πολύ συχνά το πρότυπο θεωρείται ότι είναι ειδικότερα σε διευθυντικές θέσεις, σε κέρυες επαγγελματικές θέσεις οι γυναίκες συνήθως βλέπουν ε, τους άντρες ως μοντέλα σε κάποιους επαγγελματικούς τομείς οπότε κάτι θα πρέπει να γίνει για να τα αλλάξουμε αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια και τις σκιώδεις εισηγήτριες για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η υποθεσμία καταθέσεως τροπολογιών προβλέπεται για την 25η μέχρι τέλους της εργάσιμης ημέρας. 5 ή 6 το απόγευμα κάπου εκεί. 20 Μαΐου λοιπόν έτσι για την κατάθεση τροπολογιών για την έκθεσή σας. Στα διάφορα δεν έχουμε τίποτα ώστε σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή επάνωδο στις χώρες σας.